θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Κυρίε και κύριοι, η κυρία Άνεμι Νέιτς Οτερμπουκ θα είναι ε, μέλος του Κοινοβουλίου από την 1η Πρώτου 2015 βάσει του, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Θέλω να ευχαριστήσω τον, την κυρία Ανεμή Νέιτς για το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της εύχομαι κάθε επιτυχία στο Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας της, όπου θα συνεχίσει. Οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μου ζήτησαν την άρση της ε, ασυλίας του